των Επιτροπών. Οι αλλαγές αυτές θα δημοσιευτούν στα πρακτικά. Αν δεν υπάρξει όταν γίνει έξω των πρακτικών κάποια αντίρρηση, τότε θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί αυτές οι τροποποίησεις της σύνθεσης των Επιτροπών. Από το